Il Ο πρόεδρος λέει καλημέρα σε όλους. Κύριε Σωτήνα, αρχή τη συνεδριά σα ξεκινούμε την ανακοίνωση των ε, αποτελεσμάτων. Αφορά την τέταρτη ψηφοφορία για τι τροπολογίε για το κοινό ε, ψήφισμα για την συντονισμένη δράση τη Ένωση για καταπολέμηση τη επιδημία COVID-19 και των συνεπειών τη. Όλα αυτά θα προβληθούν στην ε, οθόνη. Έχουμε την τροπολογία 53 η οποία ε, απορρίπτεται, η 54 απορρίπτεται, η 76 απορρίπτεται, η παράγραφος 43 ε, πρώτο τμήμα εγκρίνεται, παράγραφος 43 ε, δεύτερο τμήμα εγκρίνεται, ε, 48 εγκρίνεται, 77 απορρίπτεται, 24 εγκρίνεται. Παράγραφος, πριν ήταν τροπολογίες, παράγραφος 45 εγκρίνεται. Τροπολογία 18 απορρίπτεται. Τροπολογία 17 απορρίπτεται. Τροπολογία 25 εγκρίνεται. Τροπολογία 8 εγκρίνεται. Τροπολογία 9 εγκρίνεται. Τροπολογία 78 απορρίπτεται. Παράγραφος 51, πρώτο τμήμα, εγκρίνεται. Παράγραφος 51, δεύτερο τμήμα, εγκρίνεται. Παράγραφος 51, τρίτο τμήμα, εγκρίνεται. Τροπολογία 30, εγκρίνεται. Τροπολογία 1, απορρίπτεται. Παράγραφος 52 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. Παράγραφος 52 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 52 τρίτο τμήμα εγκρίνεται. 52 τέταρτο τμήμα εγκρίνεται. 53 πρώτο τμήμα εγκρίνεται. 53 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται. 55 πρώτο τμήμα εγκρίνεται 55 δεύτερο τμήμα εγκρίνεται τροπολογία 22 εγκρίνεται Ετιολογική σκέψη Β εγκρίνεται τροπολογία 31 απορρίπτεται Και τώρα προχωρούμε. Πρόκειται για την πρώτη ψηφοφορία που αφορούν ε, ε, τα συγκεκριμένα μέτρα όσον αφορά την ευελιξία για την αξιοποίηση των ε, διαρθρωτικών ταμείων. Συγκεκριμένα μέτρα για αντιμετώπιση του κορονοϊού COVID-19 στήριξη όσον αφορά την τομία, την αλία και την ε, ηχθειοκαλλιέργεια. Η ψηφοφορία θα γίνει σύμφωνα με την ίδια διαδικασία που ίσχυσε και χθες. Τώρα πια είμαστε ειδικοί και η πρώτη ψηφοφορία ξεκινάει από τώρα μέχρι τις 10 έναρξη της ψηφορίας θα ψηφίσουμε μέχρι τις 10 και τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στις 12.30. Όλες οι ψηφοφορίες πρόκειται να γίνουν ως ονομαστικές και μπορείτε να επαληθεύσετε την ψηφοφορία και τα αποτελέσματα μέσω του εγγράφου το οποίο πρόκειται να αναρτηθεί στο website της Ολομέλειας. Οπότε θα τα ξαναπούμε στις 12.30 για τα αποτελέσματα αυτής της πρώτης ψηφοφορικής. Σας ευχαριστώ. Il Presidente. Buongiorno. Ο Πρόεδρος λέει καλημέρα εις όλους. Καλώ ορίσατε. Συνεχίζεται η σύνοδος. Έχουμε τώρα το αποτέλεσμα της πρώτης ψηφοφορίας. Πρώτα-πρώτα έχουμε τις ε, τροπολογίες. 95 του 2020. Πρώτη. Τροπολογία η οποία απορρίπτεται. Τροπολογία 2 απορρίπτεται. Τροπολογία 3 απορρίπτεται. «09 του 20 η τροπολογία 3 ε, ε, απορρίπτεται, η 2 ε, εγκρίνεται, η 4 απορρίπτεται, η παριθμόν 1 εγκρίνεται. Και τώρα ψηφίζουμε. 93 του 20 όσον αφορά την ε, υδατοκαλλιέργεια. Πρώτη τροπολογία απορρίπτεται, 9 εγκρίνεται. Περιθμόν 2 απορρίπτεται. 10 εγκρίνεται. 11 εγκρίνεται. 3 απορρίπτεται. 12 εγκρίνεται. 13 εγκρίνεται. 14. Ε, εγκρίνεται. 4. Απορρίπτονται. 15. Εγκρίνεται. 5. Εγκρίνεται. 6. Εγκρίνεται. 7. Εγκρίνεται. 8. Εγκρίνεται. 16. Απορρίπτονται. Και τώρα ψηφίζουμε το 98 του 20 όσον αφορά τα ιατροτεχνολογικά. Παριθμόν 1. Εγκρίνεται. 2. Εγκρίνεται. 3. Εγκρίνεται. 4. Εγκρίνεται. 4 δέλτα σωστότερο. Και αυτά είναι τα αποτέλεσματα τη πρώτη ε, ψηφοφορία. Τώρα πάμε στη δεύτερη ψηφοφορία τη ε, σήμερα. Έχουμε τι τελικέ ψηφοφορίε. Αφορούν το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 1. Σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού αριθμό 2. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξία για το 2020. Κινητοποίηση του μηχανισμού ευελιξία για το 2020 του περιθωρίου για απρόβλεπτες ανάγκες το 20 ειδικά μέτρα για την παροχή έκτακτης ευελιξίας για την χρήση των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων. Θέσπιση ειδικών μέτρων για αντιμετώπιση της κρίσης του COVID-19. Ειδικά μέτρα ούτω ώστε να αντιμετωπιστούν τα αποτελέσματα της πανδημίας όσον αφορά την αλία και την υδατοκαλλιέργεια. Ε, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και και τέλος θα ψηφίσουμε το κοινό ψήφισμα για τη συντονισμένη δράση της Ένωσης για τα πολέμηση της πανδημίας και των συνεπειών της. Η δεύτερη ψηφοφορία ξεκινά στις 12.30. Τώρα, ουσιαστικά. Και θα διαρκέσει μέχρι τις 1.30. και Έναρξη ψηφοφορίας. Στις 4 θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα. Ευχαριστούμε και καλή συνέχεια.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 αρχά Test, test, test, test. 1, 1, 2. Voilà, test 1. OK, t'as bon son.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 Il Presidente. Grazie, buonasera. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Buonasera, Επαναλαμβάνεται η συνεδρίαση. Έχω λάβει τις θέσεις ε, του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση για τον κανονισμό που σχετίζεται για ζητήματα μετανάστευσης και διεθνούς προστασίας. Ο σχετικός κανονισμός για τις ηλεκτρονικές πληροφορίες μεταφοράς αγαθών για την μέγιστη περίοδο διακοπής ε, και ανάπαυσης ε, και για την λειτουργία των ταχογράφων. Ο κανονισμός ο οποίος τροποποιεί τους κανονισμούς 1071 και 1072 και 1024 που αφορούν την εξέλιξη των οδικών μεταφορών. Έχω λάβει επίσης την οδηγία για την ανάπαυση των οδηγών οδικών μεταφορών, τον κανονισμό για τις ελάχιστες προδιαγραφές για την χρήση νερού. Όλα αυτά βρίσκονται στα πρακτικά της σημερινή συνεδρίασης και άρα ξεκινάει από αύριο η προθεσμία τριών μηνών από τις 18 Απριλίου. Οπότε περνάμε τώρα στα αποτελέσματα του δεύτερου γύρου ψηφοφορίας. Τελική ψηφοφορία για το σχέδιο διορθωτικού προπολογισμού υπαριθμών 1. Ψήφισαν 696 591 99 υπέρ, αποχές 27, άρα εγκρίνεται με 20 ψήφους κατά τελική ψηφοφορία για το σχέδιο προπολογισμού υπαριθμών 2 ψήφισαν 696 υπέρ 691 κατά 4 αποχές μία εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας ε, ψήφισαν 696 υπέρ 603 κατά 18 αποχές 75 εγκρίνεται. Ψηφοφορία για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για το 2020 ψήφισαν 695 υπέρ 665 κατά 10 αποχές 20 εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για την κινητοποίηση του περιθωρίου για πρόβλημα γεγονότα του 2020 ψήφισαν 696 υπέρ 690 κατά τέσσερις αποχές δύο εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για τα συγκεκριμένα μέτρα για την εξαιρετική ευελιξία για την χρήση των διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων ψήφισαν 696 υπέρ 689 κατά 6 άποχες μία εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για ειδικά μέτρα για να ανταποκριθούμε στην κρίση του COVID-19 ψήφισαν 696 υπέρ 686 κατά 7 αποχές 3 εγκρίνεται τελική ψηφοφορία για τα συγκεκριμένα μέτρα για να περιοριστεί ο αντίκτυπος πανδημίας COVID-19 στο μέα αλληλείας, ηχθειοκαλλιέργειας, ψήφισαν 696 υπέρ 671 κατά 10 αποχές 15 εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για ιατρικές συσκευές 696 ψήφισαν 693 υπέρ, μία ψήφος κατά αποχές 2 εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία για την πρόταση κοινού ψηφίσματος για την κοινή αντίδραση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να πολεμήσουμε την πανδημία του COVID-19 και τις συνέπειές της. Ψηφίσαντες 694, 395 υπέρ κατά 171 αποχές 128 εγκρίνεται το ψήφισμα αυτό λοιπόν εγκρίνεται κάποιες ανακοινώσεις υπογραφή των κειμένων του διορθωτικού προϋπολογισμού υπαριθμών 2-2020 σύμφωνα με το άρθρο 97 του κανονισμού του Κοινοβουλίου. Θα ήθελα επίσης να σας ενημερώσω πως μαζί με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου θα υπογράψω δύο κείμενα για την κινητοποίηση του μέσου ευελιξίας για το 2020 και ένα κείμενο για την κινητοποίηση έκτακτων κονδυλίων. Οι σχετικοί τίτλοι θα δημοσιευτούν στα πρακτικά της σημερινής συνεδρίασης. Κλείνουμε με αυτά. Αυτά θα τα υπογράψουμε λοιπόν. Ωραία, σας ευχαριστώ. τα πρακτικά της συνεδρίασης 16ης ε, και 17ης του Κοινοβουλίου θα είναι στη διάθεσή σας στην αρχή της επόμενης συνεδρίασης. Εάν μου επιτρέπετε θα απευθύνω τα αποτελέσματα της σημερινής συνεδρίασης στους αρμόδιους φορείς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους που συμμετείχαν και είχαν την υπομονή να χρησιμοποιήσουν αυτήν την μέθοδο η οποία επιτρέπει στο Κοινοβούλιο να λειτουργεί. Είμαστε συνηθισμένοι πλέον ε, να εργαζόμαστε έτσι και είναι νομίζω και πάρα πολύ σημαντικό και για τα αποτελέσματα και βλέπουμε και τη συμμετοχή η οποία ήταν ε, αρκετά μεγάλη. Βεβαίως ε, θα ήθελα να σας ενθάρρυνω όλους να συνεχίσετε να είστε δραστήριοι στην δύσκολη αυτή στιγμή. Πριν από λίγες ε, ημέρες ε, πέθανε ένας μεγάλος ε, συγγραφέας ο οποίος θεωρούσε την Ευρώπη πατρίδα του και θα ήθελα να αφιερώσω κάποια λόγια του. Θαυμάζω όσους αντιστέκονται και δείχνουν χωρίς μεγάλες χειρονομίες ότι είναι δυνατόν να ζήσουμε, να ζήσουμε όρθιοι και στις δύσκολες στιγμές. Ο Λούις Σεπούλβεδα ένας συγγραφέας νομίζω τον οποίο έχουμε όλοι απολαύσει. Σας ευχαριστώ και καλή δουλειά.